είχα ανακοινώσει εδώ ότι ήθελα να απευθύνω ε, την πρόταση για μια νομοθετική πράξη για αλλαγή ε, ε, της οδηγίας 2016 κάθος 112 για το κοινό σύστημα του ΦΠΑ. Και το αίτημα αυτό του Ρίχαρτ Σούλικ ε, διαβάστηκε στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Η ΕΚΟΝ ε, μου είπε ότι δεν συστήνει να εγκριθεί η πρόταση αυτή. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ υπέβαλε στο κείμενο μια